Hello, colleagues. I invite you to take your seat. Χαίρετε, παρακαλώ καθίστε. Πάρτε, πάρτε τους καταλόγους ψηφοφοριών σας παρακαλώ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις κάρτες σας. για να πάει καλά η ψηφοφορία. Για να ελέγξουμε, για να μετρηθούμε. Παρακαλώ ψηφίστε ένα, μία από τις τρεις επιλογές για να μετρηθούμε. Okay. Okay. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξήντα επτά καταγεγραμμένοι. Πέρα, πέρα της ψηφοφορίας. Ωραία. Οπότε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Πρώτο θέμα, σχέδιο γνωμοδότηση για τη δεύτερη ανάγνωση, σχέδιο σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, η κυρία Κάντεμπαχ έλεγχε και δραστηριότητε που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση τη ε, νομοθεσία για τα τρόφιμα και τι ζωοτροφέ και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών τα φυτικά αναπαραγωγικά υλικά και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενιαία, μία και μόνη, άρχεται. Πέρας. Οι σοσιαλιστές έχουν μία ψήφο παραπάνω. Παρακαλώ κάποιος ε, να μην ψηφίσει. Α, ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαίρουμε την κυρία Κάντενμπαχ. Το επόμενο θέμα είναι η απαλλαγή για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης. Πρώτα απ' όλα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εισηγητής ο κύριος Λαβία. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ψηφίζουμε το τροποποιημένο σχέδιο γνωμοδότησης. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαίρουμε τον κύριο Λαβία. Επόμενη ψηφοφορία, έκθεση Λαβία. Απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το 2015. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπέρ, 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ Α, έχει αποσυρθεί. Παρά το δεν το βλέπω. Για, το, για την εύσα ψηφίζουμε, έτσι. Μα αυτό είπα ψηφίζουμε για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Δεν είπα ΕΦΣΑ, είπα Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Ο κύριος Λαβία παρακαλώ. Με συγχωρείτε, αλλά στο κατάλογο ψηφοφοριών ω σημείο 10 της μερίσιας διάταξης έχουμε την ψηφοφορία για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Αυτό ψηφίζουμε. Από την αρχή. Βεβαίως. Αλλά εγώ είπα Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Γιατί αυτό έλαβα εδώ από τη γραμματεία. Οπότε προτείνω να συνεχίσουμε την ψηφοφορία την ψηφοφορία για την ΕΦΣΑ. Γιατί αυτή ψηφίζουμε. Και θα ξανακάνουμε τις πρώτες τροπολογίες για την ΕΦΣΑ. Να ψηφίσουμε λοιπόν την ΕΦΣΑ. Α, δεν το θέλετε. Κύριε Λαβία, σας παρακαλώ, κάντε μια πρόταση. Από πλευράς μου μπορούμε να ψηφίσουμε και την ΕΦΣΑ. Αλλά έχουμε μια ημερήσια διάταξη, δεν την τροποποιήσαμε και στην ε, ημερήσια διάταξη το σημείο 10 είναι απαλλαγή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Άριστος καλύτερα λοιπόν να ψηφίσουμε με τη σωστή σειρά. Ωραία. Ωραία. Απαλλαγή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Τροπολογία 1. Υπέρ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 Τώρα ψηφίζουμε για την ΕΦΣΑ. Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Απαλλαγή 2015. Ο κύριο Λαβία είναι πάλι ο Συγητή. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές. Ξανά δεν ήταν σαφές. Υπέρ της τροπολογίας 3 παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, καλώς. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της προφορίες. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 με μια προφορική τροποποίηση των πρασίνων. Είναι κανείς κατά της προφορικής ε, τροπολογίας? Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε συνεπώς την τροπολογία με την τροποποίηση την προφορική. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Τροπολογία 17. Ψηφίστε παρακαλώ. Ε, υπέρ της απορρίφθηκε όντως. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία τώρα την τροποποιημένη γνωμοδότηση. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κύριε Λαβία. Τώρα φτάνουμε στην Εύσα. στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Απαλλαγή 2015 για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Τροπολίγα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. αποχέ Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλώς. Τροπολογία 12. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά παρακαλώ, γιατί δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 17. Υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές εγκρίνεται. 19. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Εδώ έχουμε μια προφορική τροποποίηση Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 11 με την 18, διορθώνει ο Πρόεδρος, τροπολογία 18. Υπέρ με την προφορική τροπολογία. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία, το σχέδιο τροπομένης γνωμοδότησης, ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά, πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κύριε Λαβία. Και τώρα περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία, απαλλαγή 2015 για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. ECDC. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές,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 Καλά τα καταφέραμε. Επόμενο θέμα. Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου. Ψηφίζουμε. Την πρόταση ψηφίσματος με πολλούς συντάκτες, συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στην 67 έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Α, καταπίπτει. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 76 καταπίπτει. Ναι. Ε, ψηφίζουμε την 76 τελικά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Πάλι σας παρακαλώ. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Όχι. Ξανά παρακαλώ, 97 υπέρ Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101. Άρχεται η ψηφοφορία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές υπέρ. 112 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Υπέρ, υπέρ παρακαλώ. 113. Κατά. Αποχές. Δεν έχω κάποια ένδειξη από τους σοσιαλιστές. Ας ελέγξουμε λοιπόν. 113 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται, σας ευχαριστώ. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 115. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Ας ελέγξουμε τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 14. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, είμαι πολύ τυχερή. 15. 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές. Πάλι παρακαλώ, 24 υπέρ, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Πάλι 37, 37. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 37, άρχεται ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. 38 υπέρ, 38 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές δεν ε, ε σας είδα όλους 48 υπέρ εντάξει εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50, α δεν ψηφίζουμε την 51, 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας και εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας συγχαρούμε, να συγχαρούμε τους συνεισηγητές. Το επόμενο θέμα είναι μία πρόταση γνωμοδότησης για την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η κυρία Μελά είναι η συγγήτρια. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Α, καταπίπτει.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 κατά αποχές απορρίπτεται 75 και 95 υπέρ ναι ναι 75 και 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 77 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 και 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές απορρίπτεται, 94 υπέρ, κατά, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ α καταπίπτει α έτσι αλλάζει λίγο η ρουτίνα τίποτα άλλο α όχι 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 α όχι 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 Α, πολλές καταπίπτουν. Και πάμε στην 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 66 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και να ψηφίσουμε τώρα την, την τροποποιημένη πρόταση γνωμοδότησης επειδή όμως ε, δεν εγκρίθηκε καμία τροπολογία, βασικά ψηφίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ψηφίζουμε υπέρ κατά της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης που εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής. Άρχεται. Πέρας. Οι σοσιαλιστές ε, έχουν έναν πλεονάζοντα. Περιμένουμε. Τώρα είμαστε εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε δεν έχουμε σχέδιο νομοδότησης επί της προτάσεως της Επιτροπής. Η κυρία Μελά. Κυρία Πρόεδρε, μια κουβέντα μόνο. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες και όλους τους κοιόδης που εργάστηκαν για αυτό το θέμα. Για άλλη μια φορά, όπως και για το θέμα για το οποίο ήμουν εισηγήτρια στην απασχόληση πρόσβαση στα, στη πρόσβαση στα φάρμακα που θα δούμε τώρα, όπου απορρίφθηκε η πρόταση, όχι από τους συναδέλφους, φυσικά, που πάντα θέλουν να προστατεύσουμε την υγεία και το περιβάλλον, που είναι τόσο σοβαρά θέματα έναντι της έκθεσης ε, καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες, αλλά είμαι απόλυτα ήρεμη και η ομάδα μου πιστεύω. Και θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι αποδείξαμε ότι υπάρχει ανάγκη ευρωσκεπτικισμού έναντι του τρόπου λειτουργίας ε, των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Το επόμενο θέμα. Η επόμενη ψηφοφορία που είναι σχέδιο γνωμοδότησης για την έκθεση Dorfman. Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών εν ώψη της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς. Έκθεση Ντόρφμαν. Να αρχίσουμε. Είστε έτοιμοι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Θέλετε 97 πάλι, ωραία, 97. Δυνατά τη χειρός υπέρ. Κατά. Ωραία, θα ελέγξουμε, αλλά νομίζω ότι απορρίπτεται. Ψηφίστε πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχ... Αποχές. Δεν σηκώστε τα χέρια. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 8 και 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 105 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 108. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω, αλλά μια που είναι συμβαστική καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της φοφορίες, εγκρίθηκε. Μήπως κάποιος δεν ψήφισε. Καλώς, συμβαστική 2 τώρα. Α, όχι, 109 τώρα. Υπέρ παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. 127 διορθώνει τώρα η πρόεδρος. Υπέρ παρακαλώ. 127. Στη σελίδα 8 για μένα. Λέει πρόεδρος. 127. Υπέρ της 127 κατά αποχές απορρίπτεται. 128. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 139. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. 139. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα της 139. Ψηφίστε. Πέρασε τις προφορίες. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 6. Υπέρ. Υπέρ της συμβαστικής 6. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Συμβαστική 6. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας. και απορρίφθηκε. Δεκατρία λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 13 απορρίπτεται, πιστεύω. Θέλετε να το ελέγξουμε. Καλώς. Ελέγχουμε για την τροπολογία 13. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Θα ήταν λάθος. Τροπολογία 140. Α, όχι, καταπίπτει αυτή. Και οι επόμενες καταπίπτουν. 144 λοιπόν. Υπέρ. Κατά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 Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 και 161 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ, όχι, καταπίπτει, συγγνώμη. 176 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 όχι. Καταπίπτει. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 και 22 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. και 23 ήταν μέσα. Τώρα είμαστε στην 24. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Α, όχι. Ωραία. Ποιοι είναι υπέρ τη 30. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. Όχι. 33 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές βλέπω διαφορετική πλειοψηφία, να ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε. 37. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να αλλάξουμε για 39. Ωραία. 39. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρα τις φοφορίες, Εγκρίθηκε. Σαράντα τρία τώρα, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά,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 επειδή εγκρίθηκε η 5 καταπίπτει η 60. Οπότε πάμε στην 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 και 72 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 87 καταπίπτει ή όχι, όχι. Είναι συμβατή, ναι. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 89 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 90. Αν θέλετε να ελέγξουμε για την 89, ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 89. Έχετε κάθε δικαίωμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 90 υπέρ, κατά αποχές 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε τώρα την ε, τροποποιημένη γνωμοδότηση ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας και εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Uh, we draft. Τώρα θα ψηφίσουμε τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στα Άρμακα Είναι η τελευταία ψηφοφορία. Ας συγκεντρωθούμε λοιπόν, γιατί έχουμε μακρύ κατάλογο. Λοιπόν, η κυρία Καμπεσόν Ρουΐς είναι η συγγήτρη. Υπάρχει ένα διαδικαστικό από την κυρία Ρίδ. Όταν γίνεται τέτοιος ε, θόρυβος γύρω μου είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθώ. Σας παρακαλώ, ε, θα ήταν σκόπο να μην μιλάτε τόσο δυνατά, ιδιαίτερα για αυτούς που δεν ακούν ε, πολύ καλά. Ναι, και εγώ έχω θέμα συγκέντρωσης, λέει η Πρόεδρος. Αρχίζουμε λοιπόν με τη συμβαστική 37. Υπέρ. Κατά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 κατά, αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 2, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. ΠΕΤΗ 6, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 161, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΠΕΤΗ 5, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΠΕΤΗ 26, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 165 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίφθηκε. Δεβε 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 6 στο δικό μου κατάλογο. 5.13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 και 196 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε αν θέλετε. 187 ελέγχουμε. Πέρας εγκρίνεται. Ωραία. Τροπολογία 9, συμβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβασμός 38, ε, υπέρ. Σελίδα 8, κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 8. Σελίδα 10. Συμβαστική 35, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 210. 210 Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 210. Άρχεται η ψηφοφορία. Θα ήθελα κάποια ένδειξη από τις ομάδες, εντάξει, πέρας, απορρίπτεται. 2.15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 2.15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 213 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Ας ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 214. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Και απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ωραία. Ελέγχουμε τη 216. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύε 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέτει ένα πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 529, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 39, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε, ελέγχουμε την 39. Πέρας. Ε. Και ο κύριος Τσίριο. Να ψηφίσει. Και η κυρία Αγιούσο. Αρχίζουμε και πάλι ή θέλουν να ψηφίσουν και εκείνοι. Τη στιγμή που είναι παρόντα τα μέλη δικαιούνται να ψηφίσουν. Η θέλουν να ψηφίσουν και εκείνοι. Τη στιγμή που είναι παρόντα τα μέλη, δικαιούνται να ψηφίσουν. Η κυρία Ντάλ. Νομίζω ότι είχαμε ένα προηγούμενο στην ψηφοφορία ETS και δεν ξανάρχισε η ψηφοφορία, δεν ξανά Άρα δεν πρέπει να γίνει ούτε εδώ κάτι τέτοιο. Η κυρία Γιούσο. Με μικρόφωνο. Να μην κλείνετε τόσο γρήγορα την ψηφοφορία, γιατί μόλις λέτε ότι άρχεται, λίγη κιόλας και δεν προλαβαίνουμε προχωράτε πολύ γρήγορα στη λήξη της ψηφοφορίας. Αν εξαρτάτε από εμένα, θα ξαναρχίσω την ψηφοφορία. Ξέρω ότι είναι τμηματική και θα κρατήσουμε αυτό το αποτέλεσμα τώρα και φυσικά θα επιβραδύνω στη συνέχεια. Συμβιβαστική 39. Την ψηφίσαμε, την ψηφίσαμε. Η οποία και εγκρίνεται. «280 υπέρ». «280 υπέρ». «Κατά». «Αποχές». «Εγκρίνεται». «242 και 43 υπέρ». «Κατά». «Αποχές». «Εγκρίνονται». Ζητήσατε έλεγχο για τις 2.42, 2.43, 2.45. Ας αρχίσουμε καταρχήν με τις δύο πρώτες. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Μπορώ να σας λέω ψηφίσατε όλοι. Αν θέλετε θα εισαγάγω και αυτή την πρόταση. Ωραία, πέρας. Απορρίπτεται. 247 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 248 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 244 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την 244. Άρχεται η ψηφοφορία για την 244. Πέρας. Και απορρίπτεται ισοψηφία. 246 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μα καταψηφίσατε. 246 ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 36 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 1 υπέρ. Ξεχωριστή ψηφοφορία υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 16 υπέρ Α, όχι, καταπίπτει. 254 υπέρ. Τι θέλετε να ελέγξω. Το δεύτερο τμήμα της Γιούρι 1, εντάξει. Σας παρακαλώ όμως, ε, εάν πρέπει να οπισθοδρομούμε συνέχεια, δεν γίνεται έτσι. 255. 255 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία, ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη 255. Δεν, δεν μπορώ, αν δεν βλέπω τα χέρια σας, να εικάσω ποιος ψηφίζει τι και πώς. Πέρας. Απορρίπτεται. Βασίζομαι στα χέρια που βλέπω. Δεν μπορώ να μετρήσω τις ψήφους κάθε πολιτικής ομάδας χωριστά. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ. 200... Πρέπει να ψηφίσουμε 266 και 268. Α, μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 284 και 285 από κοινού υπέρ όχι. Θέλετε να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Σύμφωνοι. Ωραία. Ψηφίζουμε ξεχωριστά. 284 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 285 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 299 καταπίπτει. Όχι, 299 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 292 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 292 άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Πέτει 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα της 296 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της 296 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 297 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Αν θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 300. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 13. Πέρας. Εγκρίνεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ να φαίνονται τα χέρια. Είμαστε στη σελίδα 26. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 532 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε, ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. 32. 5 32. Πέρας και εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει και ψηφίζουμε την 319 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. 329 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 322 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 323 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 325 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ε, κάθε φορά που λέω απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, σε ελέγξουμε. 326. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας και πράγματι απορρίπτεται με ισοψηφία. Τυχαία, τυχαία λέει η πρόεδρος. 327 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. 328 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 5-9 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 5-10 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 41 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 342 υπέρ. Κατά, αποχές Ποια ήταν η ένδειξή σα υπέρ. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 345 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 346 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 351 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 355 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 355. 355. Να ελέγξουμε. Καλύτερα ηλεκτρονικά. Ωραία. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 355. Εγκρίνεται. Εσείς χάνετε χρόνο, όχι εγώ. Εγώ θα μείνω εδώ όλη την ημέρα. Δεν βιάζομαι καθόλου. 356. 379, 361 από κοινού υπέρ. Κατά ελέγχουμε τις τρεις αυτές τροπολογίες και απορρίπτονται. 362 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ, κατά αποχές δεν βλέπω η Άλντε πώς ψήφισε. Ελέγχουμε λοιπόν γιατί δεν είχαμε σαφή ένδειξη. Ελέγχουμε λοιπόν την 363. 363. Πέρας εγκρίνεται. 364 υπέρ. Κατά. Εγώ θεωρώ ότι εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε. 364 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 380 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 537 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 378 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 390 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 404 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τετρακόσια πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 420 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 424. Νομίζω ότι εγκρίθηκε η 423. Θέλετε να ελέγξουμε. Τι θέλετε να ελέγξουμε. 424. Προχωράμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η Άλντε δεν ψήφισε υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Πρέπει να συμβαδίζουμε την κυρία Καμπεσόν γιατί είναι συγγήτρια. Πέρας. Απορρίπτεται. Είχε δίκιο. 425, 425 υπέρ κατά εγκρίνεται 427 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεβε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 436 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 449, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 451, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 468 υπέρ, κατά αποχές. Το ECR πώς ψήφισε. 468 υπέρ, κατά αποχές. Α, ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 467. Πέρας. Και απορρίπτεται. Συμβιβαστική 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίν. 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 51, ΔΕΒΕ 17, υπέρ. Στο πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα. ΔΕΒΕ 17, πρώτο τμήμα. Κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα. Α, με συγχωρείτε. ΔΕΒΕ 17, πρώτο τμήμα. Απορρίφθηκε για πληροφόρησή σας. Άρα τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 482 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 487 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Είμαι φεύγει. 488 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε στη σελίδα 54 έχουμε τη συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 503 υπέρ Όχι, όχι, μετά διαμαρτύρεστε να ψηφίζουμε από κοινού. Υπέρ τη 503 παρακαλώ. Ναι, είναι ταυτόσιμε. Ωραία. 503 κατά αποχέ εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Είναι συμβαστική βεβαίω. 514 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 516 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στη σελίδα 58, συμβαστική 45 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 553 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 554 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Α, θέλετε έλεγχο. Ωραία, ελέγχουμε την 554. Πέρας. Απορρίπτεται. Ντέβε 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 555 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 264 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 566. 566 υπέρ. Συγγνώμη, καλύτερα η 560 και η 561, όχι. Α, ωραία, σωστά λοιπόν. 566 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 567 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 568 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 569 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 523 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ελέγχουμε την 523. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 571. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 572. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 573. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Λοιπόν, δεν βλέπω ότι κάνει το ΙΣΙΑ. Παρακαλώ, 5.73 και πάλι. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5.74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5.75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έχουμε διάφορες που είναι ταυτόσιμες, αρχίζοντας με την 583. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Αν θέλετε έλεγχο, μάλιστα. Το ECR δεν μου δείχνει τι κάνει σήμερα. Πέρασε τις προφορίες. Εγκρίνεται. 588. Α, όχι. Καταπίπτει. 589. Υπέρ. 589. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 919. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 69. Τροπολογία 6.11 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας την ελέγξουμε. 6.11. 6.11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 6.12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6.14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6-15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ντεβε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι α, καταπίπτει. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ανέλεξουμε. Ελέγχουμε την 18. Άρχεται. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι. Ένας δεν ψήφισε. Πέρας. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι και εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 11. Ωραία, ας ελέγξουμε την 11. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας και εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 13. Ελέγχουμε την 13. Πέρας. Σχεδόν πέρας. Τώρα ναι. Απορρίπτεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. 32 και 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 και 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εντάξει, ωραία. Γιούρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι ε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. 83 υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, έλεγχος. Ελέγχουμε. Την 96 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 97. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 97 υπέρ. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος της 97. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 97 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι. Απορρίπτεται. Καλά απορρίπτεται. Ωραία. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 142. Δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 και η Τζούρι ε, άι, υπέρ κατά ποχές, απορρίπτονται 151 υπέρ κατά ποχές, απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο καλά. Ελέγχουμε την 154. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Γιούρι J δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε, θέλετε να ελέγξετε ακόμη και την τελευταία. Ωραία. Α, ας την ελέγξουμε και αυτή. Jury J δεύτερο τμήμα. Jury J δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Jury J δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τρεις δεν έχουν ακόμη ψηφίσει. Θα ψηφίσετε. Ε, καλά, ας κλείσουμε την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα, η τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική, άρχεται. Ένας δεν έχει ψηφίσει, μία ψήφος λείπει. Ωραία, πέρασε. εγκρίνεται. Και συγχαίρομαι ιδιαίτερα την εισηγήτρια και γενικώ όλους όσους συμμετείχαν στην πληροφορία. Και το απόγευμα θα ψηφίσουμε μαζί με την ΑΦΕΤ για τη στρατηγική μας για την Αρκτική. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη. Yeah,